άρχονται οι εργασίες της Ιλομέλειας ε, μετά την τελευταία σύνοδο στις 27 Νοεμβρίου του 2011. Έχετε λάβει τα πρακτικά. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, τότε εγκρίνονται. Θα ήθελα να κάνω διάφορες ανακοινώσεις. Σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια ομάδα ε, ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ιεμένη, την κυρία Άμαλ Μπάσα, τον κύριο Εζαντίν Αλασμπάχη και την κυρία Τάουακολ Κάρμαν που είναι δημοσιογράφος, πολιτικός και πρόεδρος της Ένωσης των ε, Γυναικών Δημοσιογράφων, αδέσμευτων γυναικών δημοσιογράφων, καθώς και συντονιστής ε, της εξέγερσης ε, των νέων στην Ιεμένη. Είναι μία από τις τρεις γυναίκες που θα λάβουν Εντό ολίγου ε, το Νομπέλ για τον μη βίαιο, ε, το Νομπέλ Ειρήνη, συγγνώμη, για τον μη βίαιο αγώνα για την ε, ασφάλεια των γυναικών και τα δικαιώματα των γυναικών. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην Τουρκία για την επίσημη επίσκεψη. Ε, Προσφώνησα το κοινοβούλιο, συναντήθηκα με εκπροσώπους